ο κύριος Βίκτορ Μανουέλ Ντασίλβα Καλτέρα. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μελή, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή για μένα να πάρω μέρος της συνάντησης αυτή σήμερα για την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2009. Την έκθεση σας παρουσίασα ήδη σε εσά κύριε Πρόεδρε και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τέσσερα βασικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Πρώτον, οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδουν μια γνήσια παρουσίαση, μια δίκαιη και γνήσια παρουσίαση των δημοσιονομικών και των αποτελεσμάτων των οικονομικών επιχειρήσεων όπως επίσης και των ε, ροών των οικονομικών.